Ε, στην ε, σχέσεις ε, της αντιπροσωπείας της Μικτής με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, συνεπώς ο διορισμός του εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της εισήγηση του κυρίου Μέρκ για την πολιτική για το ραδιοφάσμα, το ηλεκτρικό. Είναι παρόν. Ε, με συγχωρείτε. Κύριε Χακμάρκ, σας δίνω τον λόγο. Είστε εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Με την απόφαση για, το ευρωπαϊκό, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ραδιοφάσματος αναλαμβάνουμε σημαντικά βήματα προκειμένου να ανακτήσουμε τον ηγετικό ρόλο από ευρωπαϊκή σκοπιάς ε, για το ραδιοφάσμα. Υπάρχουν δυνατότητες μέσω αυτού οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ε, τηλεπικοινωνιών να έχουν νέες ευκαιρίες και φυσικά θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι όλο το νόημα αυτής της συζήτησης ε, και της απόφασης. Όχι μόνο οι τηλεπικοινωνίες, αλλά να δώσουμε νέες δυνατότητες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω, κυρία Επίτροπε, την Ουγγρική και Πολωνική Προεδρία και τους κοιόδης εισηγητές για τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Εδώ και αρκετό καιρό η Ευρώπη είχε ηγετικό ρόλο για τις ε, κινητές επικοινωνίες. Και Αυτά ήταν ε, τα κοινά πρότυπα ε, για το ευρυζωνικό δίκτυο και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία άνοιξε το δρόμο για μια ανθούσα ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία τηλεπικοινωνιών που οδήγησε σε θέσεις εργασίας και ευημερία. Δυστυχώς αυτή τη ε, νορμή τη χάσαμε. Και πλέον σήμερα ε, βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας παγκόσμιας οικονομίας με νέους παράγοντες όπως η Κίνα και η Ινδία που ανταγωνίζονται μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμάς και επομένως πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να αναλάβουμε τα ενία για το μέλλον, όχι μόνο για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών αυτών καθεαυτών, αλλά γιατί θα πρέπει να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι η ζήτηση για κίνηση ε, και μεταφορά δεδομένων ε, με, ε, μέσω κινητής τηλεφωνίας ε, αυξάνεται. Ε, μπορεί να μην εκρήγνεται, αλλά φυσικά αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχουν απαιτήσει για νέε υπηρεσίε συνεχώ. Η φιλοδοξία μου, κυρία Πρόεδρε, με την έκθεση αυτή και αυτή την απόφαση ήταν να υπάρχει ένα πολυετές πρόγραμμα ραδιοφάσματος ώστε να αναλάβουμε και πάλι τα ενία για αυτό το δεύτερο κύμα της επανάστασης του διαδικτύου την οποία βιώνουμε. Θα ήθελα να έχουμε τον ηγετικό ρόλο στη διαδικασία της αλλαγής και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες στην Ευρώπη για να έχουμε ανταγωνιστικότητα και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνονται σε θέματα τηλεπικοινωνιών. Για να σας το πω απλά, θέλω η Ευρώπη να είναι το νούμερο ένα. Όχι το νούμερο δύο, ούτε το τρία, ούτε και το τέσσερα. Αν θέλουμε όμως να βρισκόμαστε στην κορυφή, θα πρέπει να αναλάβουμε αποφάσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να βρισκόμαστε στην κορυφή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μπορέσαμε να αυξήσουμε τον πύχη ε, σε αυτή τη διαδικασία. Χάρη στην απόφαση αυτή θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τις ζώνη συχνοτήτων των 800 MHz από την 1η Ιανουαρίου του 2013, γεγονό το οποίο θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες τη δυνατότητα ε, να ε, φτάσει στο σημείο που επιθυμεί. Έτσι θα θέσουμε τους στόχους μέχρι το 2015 να έχουμε απελευθερήσει πλήρως ε, ε, τα 1200 MHz φάρματος για τη μετάδοση δεδομένων ώστε να αντιποκραθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση και ταυτόχρονα να βρισκόμαστε στην κορυφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να έχουμε τις καλύτερες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είτε είναι ο τομέας των υπηρεσιών είτε είναι ο τομέας των ε, τηλεπικοινωνιών αυτός καθεαυτών. Επίσης συμφωνήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 θα αξιολογήσει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μέτρα απελευθερωσης και άλλων συχνοτήτε, ώστε να διαφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις καλύτερες δυνατότητες. Και επίσης αποφασίσαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό αρχείο και θα διασφαλίσουμε ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες για ε, ασύρματο δίκτυο αλλά και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Με άλλα λόγια κυρία Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση η οποία θα μας δώσει δυνατότητες να επιτύχουμε ε, και να μπορέσουμε να έχουμε τον ηγετικό ρόλο στις τηλεπικοινωνίες αλλά ταυτόχρονα να αυξήσουμε και τις δυνατότητες για νέες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας και προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση και στη λήψη απόφασης αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χακμάρκ. Εξ ονόματος Επιτροπής η κυρία Κρούς θα λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πρόγραμμα ραδιοφάσματος. Όπως ξέρετε, ε, το Συμβούλιο ήδη τα αποφάσισε το Δεκέμβριο. Ελπίζω αύριο να αποφασίσει και το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή για μένα. Ε, είναι ε, ε, το, το φάσμα Γκούναρ δεν είναι ο Σπίτι Γκονζάλες επίσης οι σκιώδεις εισηγητέ ήταν μεγάλη βοήθεια και το Προεδρία. Η οθέτηση αυτού του προγράμματος θα είναι σημαντικό βήμα πρόοδου. Ξέρετε την σημασία του φάσματος για τον ψηφιακό κόσμο. Η μετάδοση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών διπλασιάζεται κάθε χρόνο με τα νέες συσκευέ στην αγορά, με την αύξηση της ζήτησης ε, και σε αυτόν τον κόσμο οι περιορισμοί στην διαθεσιμότητα του ραδιοφάσματος είναι περιορισμοί της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι δύσκολο να ε, φτάσουμε στον ε, στόχο μας χωρίς αυτήν την απόφαση, διότι θα έχουμε το 2013 θα ανοίξουμε τη συχνότητα των 800 MHz για την επόμενη γενεά. 2. Θα δημιουργήσουμε ένα αρχείο ευρωπαϊκό για να προωθήσουμε το φάσμα και το 2015 θα μπορούσαμε να έχουμε 1200 MHz. 3 ε, θα έχουμε ανταγωνιστικότητα στην χρήση του ραδιοφάσματος. Θα ε, χρειαστούμε ε, διάφορες, διάφορες άλλες, άλλα θέματα, να δούμε την προστασία των πολιτών, το περιβάλλον, το θέμα του διαδικτύου. Θα υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και θα ενισχύσουμε το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις για το ραδιοφάσμα. Και θα έχουμε στην Γενέβη την διάσκεψη είναι ένα καλό παράδειγμα και χωρίς να έχουμε αυτόν τον συμβιβασμό ε, νομίζω ε, και έχουμε επίσης τρεις δηλώσεις ε, στα πρακτικά του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις διαπραγματεύσεις στην Γενέβη. Δεν μπορώ να σας δώσω μια πλήρη αξιολόγηση παρά μόνο όταν τελειώσουν οι εργασίες. Αλλά θα καλυφθεί, θα υπάρξει μια αξιολόγηση που θα σας υποβληθεί προσεχώς. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο μου φαίνεται ότι ε, έχει ε, επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει ε, να υπάρξουν αυτές οι πρόοδοι ανάπτυξη στο ραδιοφάσμα με τον Γαλιλαίο και με διάφορες συσκευές. Επίσης ένα νέο θέμα ανεφεί στις διαπραγματεύσεις που σχετίζεται με την 700 MHz ευρυζωνικό για τις αραβικές χώρες που δεν θέλουν να περιμένουν μέχρι το 2015 για συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι λεπτό, αλλά το πρόγραμμα που συζητούμε σήμερα μας δίνει μια γραμμή πολιτικής και μέσα για εφαρμογή. Και θυμηθείτε ότι η οικονομία η μελλοντική θα είναι ψηφιακή. Μια συνεκτική πολιτική του ραδιοφάσματος θα επιτρέψει καλύτερη λειτουργία της οικονομίας για να είναι επιτυχημένη και καλό τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου να εγκρίνουν την θέση του Συμβουλίου με την απόφαση που επιτεύχθηκε τον στις 24 Οκτωβρίου πέρσι. Τώρα εξ ονόματος των ομάδων δίνω τον λόγο στον κύριο Ρούμπικ για δύο λεπτά. Και... Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ειδικά τώρα την εποχή της κρίσης, να σκεφτούμε πώς μπορούμε και πάλι να κερδίσουμε τα χρήματα τα οποία σπαταλάμε και είπατε ότι θα μετρήσουμε τα αποτελέσματα μέχρι το 2014 σημαντικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δημιουργηθούν νέες ε, προϋποθέσεις πλαίσιο που θα μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς. Και θα πρέπει να σας συγχαρώ γιατί τα πράγματα βελτιώθηκαν τα smartphones, ε, στο iPod, ε, όλα αυτά τα δίκτυα υψηλής ε, ταχύτητας που δίνουν εντελώς νέες ε, δυνατότητες και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση της ζήτησης σε αυτούς τους τομείς και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια ηγετική θέση και γι' αυτό θα ήθελα να σας συγχαρώ. Βεβαίω το ζητούμενο είναι να υπάρξουν νέες προδιαγραφές και στον τομέα του software γιατί το ζητούμενο είναι η ποιότητα, η ποσότητα, οι προτεραιότητες και οι επιδόσεις σε αυτά τα καινούρια δίκτυα. Και προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε ε, νέες τεχνικές ε, προδιαγραφές και τυποποίηση. Η Ευρώπη έδειξε ότι με νέες λύσεις software μπορεί να δημιουργήσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ε, εάν δούμε το UMT, το LT, τα δίκτυα τετάρτης γενεάς, όλα αυτά. Ποιο θα είναι το επόμενο προϊόν. Θα πρέπει να είμαστε επαρκώς προτισμένοι για μια τεράστια αύξηση του όγκου των δεδομένων. Ε, αλλά όσον αφορά την εκπαίδευση. Βλέπουμε ότι για την διαβίου μάθηση ε, όλες αυτές οι εφαρμογές είναι μεγάλη σημασίας. Επίσης τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα κοινωνικά δίκτυα, όλοι έχουν το αίτημα να έχουν πρόσβαση σε εκείνες τις συχνότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν υψηλές επιδόσεις. Η κυρία Ρέιρα Μαντουρέλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χόκμαρ και τους σκιώδεις εισηγητές, ιδίω την κυρία Τροτμάν για τα όσα έκαναν και για το γεγονός ότι συνεισέφεραν σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το πρώτο κοινό όραμα για την κατανομή του ραδιοφάσματος. Γνωρίζω ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, διότι αυτή η κατανομή του ραδιοφάσματο ε, ήταν παραδοσιακά αρμοδιότητα των κρατών μελών και μπορώ να φανταστώ πόσο περίπλοκο θα ήταν να συζητήσει το Συμβούλιο και να υπάρξουν διαπραγματεύσει για το θέμα αυτό. Υπάρχουν ε, σημαντικέ εκτεχνολογικές εξελίξει που απαιτούν νέε συχνότητε και αυτέ είναι περιορισμένε. Γι' αυτό λοιπόν η κατανομή των συχνοτήτων θα πρέπει να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο και να επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση στι πιο καινοτόμε τεχνολογίε. Η ομάδα μου χαιρετίζει τι βασικέ πτυχέ τη συμφωνίας. Ε, Μόλι μα τι υπενθύμησε η κυρία Κρό, ε, την απελευθέρωση τη ζώνη συχνοτήτων των 800 MHz για ευρυζωνικές υπηρεσίε ασημάτου διαδικτύου σε όλα τα κράτη-μέλη και από το 2013 θα πρέπει μέχρι και το 2015 να έχουμε τουλάχιστον 1.200 MHz φάσματο και επίση να υπάρχει ένα εκτενή κατάλογο των τρεχουσών χρήσεων του φάσματο για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη δυνατότητα συντονισμού και πιο αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματο. Αυτά τα μέτρα θα μα επιτρέψουν να έχουμε καλύτερε χρήσει του ραδιοφάσματο και ταυτόχρονα θα συνεισφέρουν στη μείωση του ε, ψηφιακού χάσματο. Πρόκειται για μια πρόοδο λοιπόν, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε διαδίκτυο ευρυζωνικό δίκτυο υψηλή ταχύτητα, όπω προβλέπει και η ψηφιακή ατζέντα. Και επίση θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ομάδα μου ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τη ζήτηση των ε, ε, χρηστών τηλεπικοινωνιών και τη. Ε, των όσων κατανόημουν τι ραδιοσυχνότητε για να μπορούν να ελέγχουν κατάλληλα τι συχνότητε. Στόχο μα ήταν να διασφαλώσουμε πάντα την πολιτισμική ποικιλομορφία και θεωρούμε ότι μέσω αυτή τη συμφωνία θα μπορέσουμε να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα και να προσφέρουμε εγγυώσεις στου χρήστε των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να κάνουν κατάλληλε επενδύσει σε ένα τομέα με μεγάλε δυνατότητε που θα μπορέσει να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαδουρέλ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Παναγιώτη για δύο λεπτά. Ε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που πραγματικά συνέταξε σε αυτή την ιδιαίτερως ε, σύνθετη και σημαντική έκθεση. Με την πρότασή της η Επιτροπή προτείνει να προωθήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος. Ε, αυτό πλέον είναι γεγονός, είναι τετελεσμένο. Ε, ζητούμε μια ασύρματες τηλεπικοινωνίες και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν ε, πρόσβαση στο ευρυζωνικό φάσμα μέχρι το 2012 αλλά η εναρμόνιση δεν είναι μόνο ένα τεχνικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδιαίτερως σημαντικό θέμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Μέσω της διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς και της επέκτασης στο, στην ευρυζωνικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει τις ψηφιακές δομές που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση των οικονομιών μας. Αυτή η εναρμόνιση πρόκειται να ενισχύσει τις ε, υπηρεσίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στον τομέα των υπηρεσιών. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία η οποία να εδράζεται στις γνώσεις. Διαπιστώσαμε ότι μέχρι το 2014 θα διπλασιαστεί η χρήση του ευρυζωνικού φάσματος. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτοφ. Ε, για ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Φόρτ. Ζω ότι η κίνηση όγκος θα διπλασιάζεται, θα διπλασιάζεται. Χρειαζόμαστε νέες συσκευές και ο συντονισμός ε, θα προωθήσει την ε, πρόσβαση, ε, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, καλύτερες υπηρεσίες με χαμηλότερη τιμή. Νομίζω ότι πολύ συχνά είναι ο δημόσιος τομέας που ασχολείται με το ραδιοφάσμα. Πρέπει να επελευθερωθεί και να υπάρξει ε, δυνατότητα εμπορίας ούτως ώστε να υπάρχουν νέοι πρωταγωνιστές, νέοι παίκτες. Νομίζω με το 800 MHz θα υπάρξει πρόσβαση καλύτερη και το 1200 θα δώσει καλύτερη κάλυψη στις πόλεις μας. Είναι σημαντικό να συντονιστούν οι δραστηριότητες και ε, το αρχείο κατάλογος θα βοηθήσει για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστική μας θέση οι χώρες μας θα πρέπει να απελευθερώσουν το ραδιοφάσμα. Η κατανομή, η διάθεση είναι ένα θέμα. Θα πρέπει όλοι να μπορούν να το, να το χρησιμοποιούν και χρειαζόμαστε ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές και αυτό είναι ε, καλύτερη ε, μεγάλη πρόκληση. Έχουμε μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ κυρία Φόρτ. Ε, νομίζω ότι είπατε κάτι σημαντικό, δηλαδή η διασυνοριακή ανταγωνιστικότητα. Με ενδιαφέρει να μας πείτε τι ευκαιρίες βλέπετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνή ανταγωνισμό σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείε μετά την εφαρμογή αυτής της πολιτικής ε, συχνοτήτων. Νομίζω ότι πρόκειται για την οικοδόμηση μιας υποδομής η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με τη ζήτηση. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς νομοθετούμε ε, σε σχέση με μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ε, χρειάζεται να δημιουργήσουμε κινητές υποδομές για να καταστήσουμε σύστημα ελκυστικό για τους επενδυτές. Το λόγο έχει η κυρία, ο κύριος Ζούλστρα. Η πολιτική του ραδιοφάσματος ε, συμπληρώνει την εσωτερική αγωνά. Ε, η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την, ομάδα, ε, την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε η εσωτερική αγορά, η ενή αγορά είναι η ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων αλλά και ιδεών. Δεν υπάρχουν σύνορα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών. Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων ε, έχει και κοινωνικέ διαστάσει και για την Ολλανδία. Για παράδειγμα, ξεκίνησε μία ιστοσελίδα για του πολίτε, στην οποία μπορεί κάποιο να ανταλλάξει εμπειρίε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δέκα πρέσβεις είναι κατά αυτής της δυνατότητας ε, να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους οι πολίτες. Και η Επίτροπος Κρους ε, είναι κατά της συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λανθασμένο μήνυμα που μπορούμε να αποστείλουμε στους πολίτες. Ε, το να εκφράσει κάποιο ελεύθερη την άποψή του βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατίας και αυτό είναι το μήνυμα της πολιτικής μου ομάδα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικές αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μαρσίνκεβιτς για δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που οδηγούν σε μια βελτίωση των επικοινωνιών και της μετάδοσης δεδομένων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε, αυτή την ε, τεχνολογική κούρσα, ούτως ώστε να λάβει έναν ηγετικό ρόλο ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και νομίζω ότι δεν θα πρέπει ποτέ να, δεν θα πρέπει να ε, καθυστερήσουμε όσον αφορά τη δεύτερη ανάγνωση. Η Πολωνική Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε για την έγκριση αυτής της ειδική νομοθεσίας. Επίσης η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι υπέρ της έγκρισης αυτού του κειμένου η συμφωνία να προχωρήσουμε στην ελευθέρωση της ζώνης συχνοτήτων των 800 ε, MHz για ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλες τις χώρες μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 και η επιτάχυση της ανάπτυξης κινητής ευρυζωνικότητας τουλάχιστον 300 Mbps ε, ε, και η δημιουργία ενός εκτενούς καταλόγου τρεχουσών χρήσεων του φάσματος από 400 MHz έως 6 GHz ε, θα συμβάλλει στο να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σημαντική είναι ε, η έγκριση ενός νέου ραδιοφάσματος που θα δώσει τη δυνατότητα ταχύτερης μετάδοσης δεδομένων για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα βήμα για περαιτέρω εξελίξεις και ταυτόχρονα μια εγγύηση για μια βελτίωση τη διαβίωση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Τικάου για δύο λεπτά. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, έχουμε, ε, βλέπουμε ότι θα εφαρμόσουμε το πρώτο ε, πρόγραμμα για το ραδιοφόσμα με πολιτικές και στόχους για στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της ε, χρήσης ως το 2015. Το πρόγραμμα αυτό αντανακλά τη σημασία που ε, η αποτελεσματική χρήση έχει για το, την εσωτερική αγορά της ψηφιακής επικοινωνίας και για, για την έρευνα, την ε, επιστήμη, τους δορυφορικά συστήματα, την προστασία του περιβάλλοντος, ε, της μεταφοράς κατά πολέμηση, ε, της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Νομίζω ότι στην συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περιλήφθηκαν αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να έχουμε ε, για το ένα γάμα ως στόχο να εξαλείψουμε τις ε, διακρίσεις στο ψηφιακό επίπεδο και να εξασφαλίσουμε όλοι οι πολίτες ε, να έχουν πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και να έχουμε στόχο για το 2020. Θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη ταχύτητα για την ευρυζωνικότητα και την μεγαλύτερη σύνδεση για το άρθρο 2, άρθρο 3 έχουμε τις νέες τεχνολογίες για τους καταναλωτές. Η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων πρέπει να υποστηρίζονται από τους καταναλωτές. Χαιρετίζω την συμπερίληψη στο άρθρο 4 της ανάγκης να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε ειδικό εξοπλισμό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ραδιοφάσμα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η Επιτροπή μέχρι το 2013 θα πρέπει ε, να υιοθετήσει ε, εφαρμοστικές πράξεις ούτως ώστε τα κράτη να είναι υποχρεωμένα να συλλέγουν ε, στοιχεία, δεδομένα και να έχουμε έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της απόφασης για δύο χρόνια μετά την θέση σε ισχύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Κρούς, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι περισσότεροι είναι επιφυλεκτικοί για την Ευρώπη σε αυτού του καιρού και όλοι μπορούν τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Καλό είναι λοιπόν να μπορούμε να δώσουμε και κάποια καλά νέα. Το ραδιοφάσμα είναι μια κίνηση προ ε, μια πραγματική ενιαία ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί να φοβίζει το ραδιοφέσμα, αλλά προσφέρει ε, πάμπολες δυνατότητες και μπορεί η Ευρώπη να γίνει παγκόσμιος ηγέτης σε αυτή την κοινωνία της πληροφορίας. Αυτή η συμφωνία θα ανοίξει το δρόμο για μια ανάπτυξη που θα μας βοηθήσει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην ε, ευρυζωνικότητα και στις δυνατότητές μας, στη χωροτικότητά μας. Θα μπορέσουμε να έχουμε μια ευέλικτη και συντονισμένη πολιτική ραδιοφάσματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η μεταφορά δεδομένων θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με μελλοντική ανάθεση και εισαγωγή ε, συχνοτήτων που δεν χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πανευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυστυχώς δεν μπόρεσε να επιτύχει παράταση των ε, μη αδειοδοτημένων ε, δυνατοτήτων του φάσματος για συστήματα σύρματης πρόσβασης. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε θέματα αυτά και θα πρέπει οι νέες και οι καλύτεροι τεχνολογίες να μην μειονεκτούν απλώς γιατί ήρθαν αργότερα στο προσκήνιο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νίμπλερ τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας, ο οποίος και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο υπερασπίστηκε με επιτυχία τη θέση του Κοινοβουλίου. Όλο και περισσότεροι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν κινητέ υπηρεσίε στο ίντερνετ με αυξανόμενη τάση. Το 2010 η μέση χρήση ε, από ε, διπλασιάστηκε. Ε, επίσης συνδέθηκαν πάρα πολλά iPod στο ίντερνετ και μελλοντικά θα υπάρξει μια ανωδική τάση. Η κινητή μετάδοση δεδομένων μέχρι το 2015 θα εικοσαπλασιαστεί και το 2015 780 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρησιμοποιούν ασύρματα το διαδίκτυο. Ε, γι' αυτό το ενώπιον αυτών των εξελίξεων έχει ιδιαίτερη σημασία η υπερψήφιση αυτή τη έκθεση. Θα πρέπει να μπερθούν περισσότερε συχνότητε για τι υπηρεσίε ευρυζωνικότητα, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ε, γιατί η αύξηση των συχνοτήτων ε, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τις κινητές υπηρεσίες με επιτυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν υπερψηφίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πέντε σημείων για την ευρυζωνικότητα, θα προσφέρουμε μια πολύτιμη υπηρεσία στον Ευρωπαίο πολίτη. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι μια εισηγήτρια για τον κανονισμό του roaming ε, σε σχέση με την ε, βελτίωση της ε, λειτουργίας του διαδικτύου, το οποίο θα πρέπει να γίνει πολύ φτηνότερο όσον αφορά τη χρήση του στο εξωτερικό. Και εδώ θα πρέπει να δείξετε, κύριε Επίτροπε, μεγαλύτερη τόλμη, γιατί το roaming αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και ελπίζω να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την ε, κατεύθυνση. Ο κύριος ε, Ταντζέλης για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα και ένα φιλόδοξο σχέδιο. Να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε παγκόσμιο ηγήτη σε θέματα ταχύτητας, κινητικότητας, κάλυψης και ευρυζωνικών ταχυτήτων. Ο στόχος, όπως υπενθυμίστηκε εδώ, είναι να υπάρχει ευρυζωνικό δίκτυο για όλους. Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα έχουν ήδη σε μεγάλο τμήμα του ραδιοφάσματός τους και επομένως είναι ευπρόσδεκτη η πρόθεση να απολευθερώσουμε τη ραδιοσυχνότητα των 800 MHz για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες ασύρμα διαδικτύου μέχρι τα τέλη του έτους και ευπρόσδεκτη η περαιτέρω ανάπτυξη της ταχύτητας ε, της ε, ε, μετάδοσης δεδομένων ε, με πάνω από ένα μεγαμπάιτ ανά δευτερόλεπτο. Πρόκειται για σημαντικούς στόχους. Η ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν αναπτύσσεται, ε, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και σκληρή δουλειά. Θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί προκειμένου να αναλάβουμε και πάλι τα ενία στην παγκόσμια οικονομία της πληροφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καμερεβέρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να βάλω λίγο νερό στο κρασί το οποίο δορίζεται εδώ, γιατί από πολιστική άποψη η κοινή θέση του Συμβουλίου είναι μάλλον απογοητευτική και δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Οι συχνότητες είναι ένα σπάνιο αγαθό που έχει μεγάλη πολιτιστική σημασία όσον αφορά όσο χρειάζεται το ραδιόφωνο κάποιε συχνότητε για να μεταδίδει τα προγράμματά του και να φτάνει στον πολίτη, οι συχνότητε είναι μεγάλη σημασία. Ε, έχουν γίνει εδώ ε, η Επιτροπή Πολιτισμού συγγνώμη, έκανε πολλές ε, προτάσεις για να ληφθεί ιδιαίτερος υπόψη ο ρόλος του ραδιοφώνου. Ε, είχαμε ζητήσει να υπάρχουν ξεκάθαροι αντισταθμιστικοί κανόνες για να μην δημιουργηθεί αύξηση του κόστους στα θέατρα και να εξασθεί το θέμα του, των ψηφιακών μερισμάτων. Ωστόσο, δεν ε, επιτεύχθηκαν σημαντικές ε, βελτιώσεις παρά μόνο πενιχρά αποτελέσματα. Αναμένω από τις χώρες ε, μέλη να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους και να μην κινηθούν μόνο ε, στην κατεύθυνση της ε, οικονομικής ε, σκοπιμότητας, αλλά να αναγνωρίσουν ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τις ανάγκες της πολυπολιτισμικότητας. Θα ήθελα να ζητήσω να τηρήσετε τα χρονικά σας περιθώρια και, να... και δίδω το λόγο στην κυρία Καρόλα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κούναρ Χόκμακ για την εξαίρετη εργασία σχετικά με το ραδιοφάσμα. Ε, Βεβαίω, το ραδιοφάσμα είναι πάρα πολύ περιορισμένο, το χρειαζόμαστε σε πάρα πολλούς τομείς, κυρίως ε, για την ψηφιακή τεχνολογία και τις συνδέσεις ευρυζωνικότητας. Ε, είμαι στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για το πρόγραμμα αυτό και χαίρομαι που το κείμενο είναι φιλόδοξο και σκέπτεται το μέλλον. Η ψηφιακή ατζέντα είναι και για τις απομακρυσμένες περιοχές και η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων ε, χρειάζεται ε, περαιτέρω συχνότητα ραδιοφάσματος. Τα 800 MHz ε, θα πρέπει να απελευθερωθούν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και αυτό είναι μεγάλη πρόοδος διότι ε, μερικές χώρες έχουν καθυστέρηση. Πρόκειται για φιλόδοξο επίτευγμα και νέες υπηρεσίες θα υπάρξουν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μπασόσκου, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη χρειάζεται μία ευέλικτη και συντονισμένη πολιτική για το ραδιοφάσμα. Αυτό θα πρέπει να συνεισφέρει στη συνέχεια στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Το ραδιοφάσμα είναι ικανή και αναγκαία συγχυθήκη για μια ψηφιακή κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει παγκόσμιο ηγήτη για τι ε, ταχύτητε ε, σύνδεση, την κάλυψη ε, και τι δυνατότητε του ευρυζωνικού δικτύου. Θα πρέπει να μειώσουμε τι διαφορέ μεταξύ ψηφιακών θεμάτων και θα πρέπει να επεκτείνουμε την ε, ε σε μια διαδοτημένου φάσματος για συστήματα σύρματης πρόσβασης. Η τεχνολογία αυτή θα πρέπει να είναι προσιτή και να είναι και προσβάσιμη σε ε, περιοχές της υπαίθρου και όχι μόνο σε αστικές περιοχές. Θα πρέπει επίσης να επιστήσω την προσοχή σας και στα μέτρα προστασίας κατά των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η χρήση του ραδιοφάσματος δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, γι' αυτό είναι απαραίτητο λοιπόν να παρακολουθείτε μονίμως η χρήση του ραδιοφάσματος. Ο κύριος Μάτουλα για η e, e, e χρήση του ραδιοφάσματος ε, είναι πάρα πολύ ε, σημαντική αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη για τους τελικούς δικαιούχους ε, και τους ιδιωτικούς οργανισμούς και παράγοντες. Υπάρχει βούληση των ευρωπαϊκών οργάνων να αναλάβουν πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλύτερης ταχύτητες και εναρμόνιση των συχνοτήτων στα 800 MHz. Όλα αυτά θα μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του ψηφιακού χάσματος, διότι οι μελέτες έχουν καταδείξει ότι η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό χρειαζόμαστε εναρμόνιση πολλών ζωνών. Αυτή η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποτελέσει την βάση για αύξηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας που θα μας βοηθήσει να ε, επιτύχουμε τους στόχους μας. Ε, κυρία Ζούμπα, ένα λεπτό. Οι συχνότητες του ραδιοφάσματος είναι κάτι το οποίο συζητιέται και θα πρέπει να αποφασιστεί. Οι συχνότητες για τους χρήστες των τηλεπενικοινών χρειάζονται και κάποια εποπτεία. Ε, υπάρχουν εδώ κάπως αποκλίνουσες ε, απόψεις και θα ήθελα να ακούσω σχετικά την ε, άποψη της Επιτροπής. Οι συχνότητες θα πρέπει να ανοίξουν στο κοινό και θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, επίσης για λόγους ασφάλειας, άμυνας κλπ. Και ε, θα δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα για τους ε, χρήστες. Θα απελευθερωθούν ε, ασύρματες υπηρεσίες σε διάφορες αγορές και θα ήθελα να μας δώσει σχετικά μια απάντηση κυρία Κράους ο κύριος Πάσκα, όσον αφορά τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συνοδευτικά μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2010 είχε υποβάλει πρόταση για το πολιτέ πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο του 2011 άλλαξε τους στόχους προκειμένου να δοθούν νέε δυνατότητε για να δίνονται οι κατάλληλε συχνότητε ραδιοφάσματο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ευρυζωνικά δίκτυα. Βέβαια, όλε οι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έγιναν κατανοητέ και δεν υποστηρίχθηκαν από το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και να υπάρχει αγαστό κλίμα συνεργασία. Από το 2013 και μετά, όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξουν τη ζώνη συχνοτήτων των 800 MHz και από το 2015 και τούδε θα έχουμε και τα 1200 MHz φάσματο για μετάδοση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών. Αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να διευρύνει τις ευρωπαϊκές ευρυζωνικές της συνδέσεις και να οδηγήσει σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων χρηστών. Ας ελπίσουμε πραγματικά λοιπόν να επιφέρει τα αποτελέσματα που ε, αναμένουμε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Κούναρ γιατί πραγματικά έθεσε τα θεμέλια για μια ανταγωνιστική Ευρώπη και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο το εξή. Μέχρι το 2014 ε, βάλατε ε, το στόχο... Madame Cruz, je vous parole για την απελευθέρωση της ε, ζώνης των συχνοτήτων. Ολοκληρώθηκε το Catch the κυρία Κρούς, για ε, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ένα-δυο θέματα δημιουργούν ανησυχία και μια συγκεκριμένη παρατήρηση που ακούσαμε από την κυρία Μπασέσκου και την κυρία Χάρκ που μιλούσε για την ε, ε χωρίσεις μία διαδοτημένου φάσματος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία και θα το εξετάσουμε. Επίσης αυτό συνδέεται και με τις παρατηρήσεις ε, που ακούσαμε από την κυρία Σούμπερ η δημόσια πρόσβαση θα ε, καθορίζεται από, την, από το δημιουργία του εκτενούς καταλόγου, αλλά το πάντα δεν είναι θέμα ε, εμπορίου και μόνο. Θα ήθελα να πω λοιπόν εν κατακλείδη ότι όλα τα μέλη συμφωνούν, επιτρέψτε μου να ε, κάνω αυτή την εικασία, ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, διότι αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε ανάπτυξη και θα δώσουμε μια νέα όθηση για δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνούμε όλοι από αυτού του ζητήματος, ότι ο ρόλος του ραδιοφάσματος ε, πραγματικά δίνει όθηση για ανάπτυξη στην Ευρώπη και πραγματικά έχει χειροπιαστά ωφέλη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και ότι το πρόγραμμα του ραδιοφάσματος, το οποίο θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο αύριο, θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο ότι μετά από σκληρή δουλειά από πλευράς Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είχαμε αποτέλεσμα, αλλά είναι και ένα από αυτά τα στοιχεία όπου μπορούμε να αποδείξουμε στον έξω κόσμο ότι υπάρχουν και θετικά μηνύματα και ε, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους για την επικοδομητική σας συνεργασία και για το έργο σας στη διάρκεια όλων των διαδικασών. Ε, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, αλλά Πραγματικά ε, χύθηκαν πολλά δάκρυα για το θέμα αυτό. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι το καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι έκαναν εξαιρετικά, ε, εξαιρετική δουλειά όλοι. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά για την τελευταία λέξη. Κυρία Πρόεδρε, το ραδιοφάσμα είναι περιορισμένο. Ωστόσο, οι ευκαιρίε είναι περιόριστες. Και όπως ε, είδαμε στι ε, πρόσφατε εξελίξει και όπω θα δούμε και μελλοντικά σε εξελίξεις που αντιμετωπίζουμε τώρα και νομίζω ότι είναι έντιμο να πούμε ότι ο πολιτισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα έχει περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ για να φτάσει στον ε, κοινό. Όπως βλέπετε τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία και νομίζω ότι ο πιο σημαντικός στοχασμός στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης ήταν ότι είδαμε τελευταία δεκαετία ραγδαίες εξελίξεις. Θα δούμε θα εξίσου ραγδαίες εξελίξεις την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την πλήρη χωρητικότητα για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε στο μέγιστο με νέες υπηρεσίες και είναι επίσης σημαντικό σε σχέση με τα επόμενα βήματα να εξασφαλίσουμε την ταχεία εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, αλλά ταυτόχρονα να ετοιμαστούμε για τα επόμενα βήματα. Διότι είδαμε μόνο την αρχή, την αρχή μιας νέας εξέλιξης, ενός νέου τρόπου, μιας νέας διαδικτυακής επανάστασης θα έχουμε συνέπειες και δυνατότητες, ευκαιρίες όπως είδαμε στη Βόρεια Αφρική που είδαμε με τις ε, διαμαρτυρίες όπως είχαμε την επανάσταση ε, διαφόρων τμήματων των οικονομιών μας θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα επόμενα βήματα ε, περισσότερο αν είμαστε ταχύτατοι Έχουμε ε, τα 1200 MHz στόχο για το 2015 και μετά θα υπάρχει ανάγκη να αξιολογήσουμε τις ανάγκες ε, και να προχωρήσουμε ταχύτατα τα επόμενα χρόνια ε, διότι ο χρόνος τρέχει και θα πρέπει να είμαστε επικεφαλής, να έχουμε ηγετικό ρόλο, να τον αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο και να είμαστε ο νούμερο ένα για να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες, να ανοίγουμε νέες ευκαιρίες συνεχώς, διότι είναι απεριόριστες, ενώ ε, τα μέσα, οι πόροι είναι περιορισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε ένα διαδικαστικό, κύριε Ρουμπίγκ. Κυρία... Πρόεδρε, το, μικρόφωνο, το δικό μου μικρόφωνο λειτουργεί και οι συχνότητες εδώ επίσης αλλά το κουμπί στο μικρόφωνο μου έχει χαλάσει και ζήτησα, παρακάλεσα δύο φορές να έρθει εδώ ένας τεχνικός και να διορθώσει το κουμπί αυτό. Και παρακαλώ να διορθωθεί αυτό μέχρι αύριο. Ε, θα γίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε, ευχαριστούμε όλους ε, και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30.